Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past three already. Um, ε, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε γιατί είναι ήδη 3 και 4. Ε, και θεωρώ πως τα μέλη εδώ, τα υπόλοιπα της ε, Επιτροπής ΕΡΕΚΙ θα επιστρέψουν. Ίσως επειδή είχαμε και την πρωινή συνεδρίαση, δεν έχουμε τόσα μέλη αυτή τη στιγμή μαζί μας. Ας περάσουμε όμως στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης, λοιπόν που είναι μία μελέτη που ανατέθηκε από το θεματικό τμήμα Ζ με θέμα τη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την πολιτική συνοχή. Η Ρέτζη λοιπόν ζήτησε από το θεματικό τμήμα Β να συντάξει μια τέτοια μελέτη για τη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς οι λεπτομερείς διατάξεις για αυτές τις ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της PPP περιλήφθηκε στο την τελευταία περίοδο και υπάρχει τώρα όλο ένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτήν τη δυνατότητα συνδυασμού δηλαδή κονδυλίων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τα περισσότερε από αυτέ τι συμπράξει ε, PPP εστιάστηκαν κυρίω ε, στον τομέα των ε, μεταφορών. Οπότε ορισμένα από τα πορίσματα αυτή τη μελέτη θα είναι θα σχετίζονται και με τη δική μας έκδοση εφαρμογής της πολιτικής για, τον, ε, για, τη, τις βιώσιμες μεταφορές, ε, όπου έχουμε ως εισηγητή τον κύριο Νοβάκοφ, ο οποίος παρευρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Ε, το έγγραφο λοιπόν θα παρουσιαστεί από την επικεφαλής αυτού του ερευνητικού έργου, την κυρία Λάουρα Ντελπόντε, από το Κέντρο Βιομηχανικών Μελετών του Μιλάνου. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο για αυτή την παρουσίαση και είμαστε σίγουροι ότι στο ίδιο μεταξύ θα καταφτάσουν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Να σας πω ότι χαίρομαι για το γεγονό ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τα πορίσματα αυτής της μελέτης σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την πολιτική συνοχή. Ε, αυτή λοιπόν η ε, μελέτη εξετάζει τη συλλογιστική για αυτή την ε, χρήση ε, των, των PPP και της πολιτικής συνοχής και βασίζεται σε ένα συνδυασμό από διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους, δηλαδή μια αναθεώρηση ή μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνεντεύξεις με εκπροσώπους από βασικά θεσμικά όργανα και 8 περιπτωσιολογικές μελέτες τι είναι τώρα μια PPP, μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν διαφορετικές, ε, διαφορετικοί ορισμοί γιατί υπάρχουν διαφορετικές μορφές PPP, διαφορετικές δηλαδή συμφωνίες PPP και εξαρτώνται ακριβώς από τις ε, διαφορετικές σχέσεις, ε, τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η PPP, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αποτελεί έναν γενικότερο όρο στον οποίο μπορούν να υπάγονται διαφορετικού είδους συμπράξεις. Αν μπορεί να γίνεται δηλαδή ένα outsourcing των υπηρεσιών, ε, μέχρι και να μπορεί να περιλαμβάνει μια ιδιωτικοποίηση περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου. Πάντω σε γενικέ γραμμέ αναφέρεται σε κάποιο, ε, ένα είδο συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι πιο, ε, ορισμοί, για παράδειγμα όπω αυτό που χρησιμοποιείται από το. Ε, Κέντρο Ευρωπαϊκής Ε, Με βάση λοιπόν αυτόν τον ορισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, τμήματα ε, κατασκευαστικά και διαχειριστικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα, τις συμβάσεις των PPPs, ε, θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Καταρχήν, ε, δημιουργούν ε, ή εδραιώνουν μία μακροχρόνια σχέση. Για παράδειγμα, συνήθως έχουν βάθος χρόνου 20 έως 30 ετών και επίσης βασίζονται στην απόδοση. Δηλαδή, με αυτές οι συμβάσεις εστιάζουν στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και όχι στο τι χρειάζονται ως κονδυλία. Επίσης, η κατανομή των ε, κινδύνων ε, αποτελεί έναν όρο που πάντα εμφανίζεται στις συμβάσεις, ε, δηλαδή με βάση αυτές τις PPP ο κάθε συμβαλόμενο μέρος αναλαμβάνει τους τομείς εκείνους τους οποίους θα πρέπει να είναι, είναι πιο ενδεδειγμένο να αναλάβει. Επίσης, η κλίμακα και η περιπλοκότητα είναι βασικές διαστάσεις, καθώς λαμβάνουν υπόψη τι διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωή του έργου. Ε, και ε, τέλος τα δύο τελευταία στοιχεία, δηλαδή η σχέση κόστους αποτελέσματος ε, και η δημοσιονομική διαχείριση είναι, δεν είναι πάντοτε τμήμα αυτών των συμβάσεων PPP, αλλά είναι σημαντικές έννοιες στο πλαίσιο της σύναψης τέτοιων συμφωνιών. Αυτό το value for money, δηλαδή η σχέση κόστος αποτελέσματος, είναι να αξιοποιούνται με το καλύτερο δυνατό οι δαπάνες. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πάντοτε στο πλαίσιο της σύνταξης των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη και αυτή η διάσταση. Mm. Επίσης, η δημοσιονομική τώρα μεταχείριση των δαπανών στο πλαίσιο μια PPP αποτελεί ένα διαφιλονικόμενο ζήτημα, ένα αμφισβητούμενο ζήτημα, γιατί στο πλαίσιο ε, των όσων προβλέπει σήμερα η Eurostat, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένε ε, προποθέσει μπορούν ορισμένες ε, δαπάνε PPP να περιληφθούν στου ισολογισμούς των δημοσίων επιχειρήσεων. Με αποτέλεσμα αυτό να σημαίνει ότι ουσιαστικά κάποιε υποχρεώσει του δημοσίου μετατίθενται για το μέλλον. Τώρα, ποια είναι τα δυνητικά ωφέλη αλλά και οι κίνδυνοι των PPPs. Θα πρέπει να σας πω ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι πολύ αμφιλεγόμενος και στο πολιτικό επίπεδο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και η σχετική συζήτηση παραμένει πολύ πολλωμένη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ε, πραγματικά οριστικές, ε, οριστικά τεκμήρια ή ενδείξεις ότι δηλαδή είναι υψηλότερη η απόδοση όταν χρησιμοποιούνται PPP. Δηλαδή τα αποτελέσματα των PPP εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Τα σημαντικά πάντως ωφέλη της προσέγγισης με βάση τις συμπράξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι καταρχήν η δυνατότητα αξιοποίησης, καλύτερης αξιοποίησης των δημοσίων κονδυλίων μέσω της προσέγγισης ιδιωτικών κονδυλίων και επίσης η ε, διάθεση συμπληρωματικών ακριβώς ε, ιδιωτικών ε, ε, κονδυλίων. Επίσης υπάρχουν και χαμηλότερα κόστη διαχείρισης και συντήρησης. Αντιθέτως η κίνδυνη είναι ο υψηλότερος κίνδυνος χρηματοδότησης, υψηλότερο κόστος συναλλαγός και προβλήματα που σχετίζονται με λιγότερη διαφάνεια και λιγότερη ανάληψη ευθυνών. Επίσης υπάρχει και χαμηλότερη ευελιξία η οποία σχετίζεται ακριβώς με το μεγάλο βάθος χρόνου που έχουν συνήθως οι PPP. Τώρα, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ε, των ε, αγορών PPP στην Ευρώπη. Οι σχετικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2006 αυξάνονταν σημαντικά, ε, ενώ από εκεί και μετά επλήγει σημαντικά η αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης και τότε άρχισε μια φθήνουσα πορεία. Γεωγραφικά παρατηρούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι με μεγάλη διαφορά η μεγαλύτερη αγορά για PPP στην Ευρώπη και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές PPP στον κόσμο σε ό,τι αφορά δηλαδή τον όγκο των επενδύσεων για την περίοδο 2000-2015 το 45% ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες μεγάλες αγορές είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τις PPPs, κυρίως εστιάζονται στον τομέα των μεταφορών, ειδικότερα στις, ε, στις, ε, στον οδικό τομέα. Για παράδειγμα, αντιστοιχούσε στο 56% των συνολικών PPP. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την κλίμακα, το μέγεθος των ε, έργων που ε, χρηματοδοτούνται μέσω PPPs, έχει αρχίσει να υπάρχει μείωση του ενδιαφέροντος για πολύ μεγάλα project και έχει αρχίσει τώρα τελευταία να εμφανίζεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικότερα στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υποεθνικό επίπεδο, δηλαδή περιφερειακό, για μικρή κλίμακα PPPs. Τώρα, τι έχει ε, οδηγήσει στην αυξημένη χρήση των PPP στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ακριβώς ε, η ενσωμάτωση μέσα στις ε, πολιτικές επενδύσεων του Δημοσίου, δηλαδή για την συμπλήρωση των κενών χρηματοδότησης των υποδομών. Η προσέγγιση λοιπόν ε, με βάση την πολιτική συνοχή βασίζεται ακριβώ σε αυτό το σκεπτικό, δηλαδή στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τα υψηλότερα κριτήρια σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την εστίαση στα αποτελέσματα. Στην αρχή ο συνδυασμό αυτών των δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων γινόταν σε περιπτώσει ad hoc όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της, ε, στο αεροδρόμιο της και της Λισαβόνας. Μετά από την περίοδο του 2003 άρχισε να χρησιμοποιείται ε, πιο συστηματικά και να αναφέρεται συγκεκριμένα ε, ως στόχος η αυξημένη αξιοποίηση των PPPs. Ωστόσο, μόνο στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένε διατάξει σε ό,τι αφορά αυτέ τι PPPs. Και αυτέ οι διατάξει προβλέφθηκαν έτσι ώστε να ε, μην υπάρχουν πλέον τα διοικητικού χαρακτήρα εμπόδια τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τη χρήση των PPPs. Ειδικότερα δηλαδή ο νομοθέτη έχει αναγνωρίσει ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση ε, των ευρωπαϊκών επενδυτικών και διαρθρωτικών ταμείων για ε, την υποστήριξη μέσω PPPs θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των PPPs. Άρα λοιπόν ο κανονισμό περί κοινών διατάξεων έχει επιτρέψει ακριβώ την καλύτερη ευθυγράμμιση των διαδικασιών των Grand Application και των διαδικασιών για την ε, δημοσίων συμβάσεων για αυτέ τι PPPs. Τώρα, πώ έχουν αξιοποιηθεί οι PPPs στις, ε, στην πολιτική συνοχή. Στην αρχή χρησιμοποιούνταν πολύ σποραδικά, χωρί να λαμβάνονται υπόψη στρατηγικού χαρακτήρα σκέψη, δηλαδή εστιάζονταν κυρίω σε, σε μεγάλα έργα υποδομή, ειδικότερα στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Πορτογαλία. και κυρίως εδώ εστιαζόταν σε πολύ μεγάλα έργα και βασιζόταν σε ε, μείζων σημασία σε ε, χρηματοδοτικά εργαλεία. Θεωρούμε ε, τώρα πως με την αυξημένη χρήση των ταμείων θα υπάρξει και περισσότερη σύνθετη χρήση PPP και χρηματοδοτήσεων από τα διάφορα ταμεία. Δεν υπάρχει όμως σχέση μεταξύ του επίπεδου ανάπτυξης των εθνικών αργολών PPP και της ένταξη των PPP στην πολιτική συνοχή. Και εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί ε, συμβαίνει. Γιατί οι PPP μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικέ προτεραιότητε στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματο για τι PPP, ενώ διαφορετικέ μπορεί να είναι προτεραιότητε στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή όπου εντάσσονται οι PPP. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν ε, βλέπουμε να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, διατάξεις σε ό,τι αφορά τις ε, PPPs οι οποίες ε, να καταδεικνύουν ότι πράγματι οι PPPs επιφέρουν περισσότερα αποτελέσματα. Ε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου και είναι και πολύ περιορισμένα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένο το οποίο να μας καταδεικνύει το πώς γίνεται η συνδυαστική χρήση των PPPs και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Άρα λοιπόν τα σχετικά δεδομένα δεν είναι ε, πλήρη και αφορούν μόνο μεγάλα έργα ε, τα οποία εκτελέστηκαν κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013. Όμως, εκείνο το πιο σημαντικό δηλαδή που μας λένε τα δεδομένα είναι ότι η χρήση των PPP στην πολιτική ε, συνοχή είναι πολύ περιορισμένη. Από δηλαδή από χίλια συνολικά μεγάλα έργα, μόνο τα 27 θεωρήθηκαν ως PPP. Ε, και επίσης ε, αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι εδώ ο χώρος των μεταφορών αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη. Και επίσης τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η εμπειρία σε ό,τι αφορά τη συνδυασμένη χρήση PPP και ε, χρηματοδοτικών εργαλείων εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία ποια ε, διδάγματα τώρα μπορούμε να αντλήσουμε από την εφαρμογή αυτής της, αυτών των μεικτού χαρακτήρα έργων PVP. Υπάρχουν δύο βασικοί κινητήρες δυνάμεις, αν θέλετε, ότι ε, καταρχήν εφαρμογή με τις, ε, με τις μικρότερες ε, όσο γίνεται καθυστερήσεις και υποστήριξη των δημοσίων κοντιλίων με τα ιδιωτικά. θεωρούμε πως η ε, μη ύπαρξη καταλλήλων πόρων χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο περιόρισαν τη χρήση των PPPs. Και ακριβώς και γι' αυτό δεν αξιοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό και τα σχετικά ταμεία όπως ο ERDF ε, για ε, την αξιοποίηση συνδυαστικά με τα PPPs. Και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η ψηλότερη χρήση, η πιο εκτεταμένη χρήση των PPPs οδηγεί σε υψηλότερη απορρόφηση των σχετικών χρηματοδοτικών κονδυλίων. Αντιθέτως, ορισμένες αρχές οι οποίες ε, επιθυμούν να προβούν σε μια συγχρηματοδότηση ε, μπορούν να βρίσκουν τόσο περίπλοκο το χαρακτήρα των PPP που να μην επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν. Πάντως, τα έργα τα οποία εκτελούνται με PPP συνήθως εκτελούνται και εγκαίρως και στα πλαίσια του αρχικού προϋπολογισμού. αλλά σε μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα είναι πιο μεικτού χαρακτήρα. Δηλαδή κάποια έργα τα οποία αρχικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχή σε ό,τι αφορά τις PPPs τελικά μπορούν να έχουν αρνητικές ε, οικονομικές επιπτώσεις όπως αυτό συνέβη για παράδειγμα με την γέφυρα Τάγκου στη Λισαβόνα όπου η επανειλημμένη επαναδιαπραγμάτευση μία σειρά από ε, PPPs οδήγησε σε αρνητικέ δημοσιονομικέ επιπτώσει. Ο συνδυασμό των PPPs και των πόρων από την πολιτική συνοχή μπορεί να επιφέρει ε, θετικά αποτελέσματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί, για παράδειγμα, να διασφαλιστεί η πλήρωση υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων ή η καλύτερη ένταξη κοινωνικών διαστάσεων σε έργα PPP. όλα πάντως τα PPP ε, τα οποία περιλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη κατέδειξαν ότι και οι ικανότητε αλλά και η πολιτική βούληση από την πλευρά του δημοσίου τομέα ε, ήταν εξαιρετικά σημαντικέ για την επιτυχία του. Ειδικότερα δηλαδή η δυνατότητα του δημοσίου φορέα να συντονίζει τον κύκλο ε, του έργου με τον κύκλο έργων του ERDF έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία των, ε, του, του κάθε έργου. Και αυτό επιτέθηκε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μέσω της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών για παράδειγμα, για την κατασκευή του αερολιμένα των Αθηνών, η αθηναϊκή κυβέρνηση έπρεπε να διασφαλίσει την πολύ καλή ποιότητα οδική πρόσβαση στο αερολιμένα μέχρι να, ή πριν την ολοκλήρωση τη κατασκευή του αεροδρομίου. Ή για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα έργο υποδομή ε, στην Κορνουάλη, η κυβέρνηση χρειάστηκε να διασφαλίσει καταρχήν τη μεγάλη διείσδυση ε, της σύνδεσης broadband στο διαδίκτυο για τους ε, ε κατοίκους. Οπότε ε, δεν έχουμε πολλά παραδείγματα, αλλά υπάρχουν ε, κάποιες ε, περιπτώσεις αποτυχίας των PPP, όπως για παράδειγμα εκείνο στο BRS όπου χρειάστηκε να τερματιστεί αυτή η σύμβαση PPP επειδή δεν υπήρχε ούτε πολιτική υποστήριξη αλλά και επειδή έγιναν λάθη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το βασικό αρχικό προπολογισμό. Τώρα, τι έχουν κάνει ε, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ώστε να υποστηρίξουν την αυξημένη χρήση των PPP στην πολιτική συνοχή. Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει παίξει ένα ρόλο κλειδί στην προώθηση τη χρήση γενικότερα των PPPs. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει παράσχει υποστήριξη μέσω δύο κυρίω εργαλείων. Καταρχήν, παρέχει μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν ε, έργα PPPs, δημιουργώντας δηλαδή πιο ευνοϊκές συνθήκες για τους ιδιωτικούς επενδυτές. Και τέτοιου είδους παραδείγματα μπορούν, ε, μπορούμε να αναφέρουμε το ε, Jessica και το Marketing Fund. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει και κάποιες συμβουλευτικές επιχειρήσεις αλλά δεν παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των έργων που αξιοποιούν PPPs. Σε, τώρα, στα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, μονάδες ε, κεντρικές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ε, PPPs αλλά επειδή έχουν ακριβώς περιορισμένο αριθμό δεν επιτυχάνουν να ε, ε, αποτελεσματικά τον στόχο αυτό της ε, προώθησης του συνδυασμού PPP με τα ταμεία, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η μόνη εξαίρεση είναι η Ελλάδα η οποία έχει καταφέρει να συμπεριλάβει αυτό το συνδυασμό στο προγραμματισμό της. Δύο ακόμα χώρες οι οποίες έχουν προωθήσει και αυτές την συνδυασμό των PPP με την πολιτική συνοχής είναι η Κροατία και η Πολωνία τι μπορεί τώρα να βελτιωθεί. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συμπράξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι μόνο μία από τις διάφορες εναλλακτικέ που υφίστανται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Άρα λοιπόν η χρήση των PPP θα πρέπει να βασίζεται σε μία ανάλυση της σχέσης κόστους αποτελέσματος. Επίσης αυτές οι αναλύσεις σχέσεις κόστου αποτελέσματο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τακτικά, συστηματικά από τι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα. Επίση, το μοντέλο των PPP θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα ε, στον σχεδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια ε, επενδυτικά ε, στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών που θα μπορούν να ενσωματώνονται στα διάφορα περιφερειακά προγράμματα. Επίσης, τα ωφέλη της χρήσης των PPPs στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής δεν είναι ακόμα σίγουρα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων PPP για να διαπιστωθεί και, ακόμα είναι σημαντικό να υπάρξει περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη, να αναπτυχθεί εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τα PPP τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτά ε, από την πλευρά μου παρουσίαση και αναμένουμε ενδιαφέρον τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πληρέστατη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Οπότε τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις από πλευράς των μελών της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεως. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Οι κυρίες πρώτα, ως ήθιστε. Η κυρία Νταμάτου. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των συναδέλφων που απουσιάζουν. Ποια ερώτηση είχανε. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα. Παραδείγματα μικρών έργων, μικρομεσών επιχειρήσεων που συνέβαλαν κατά κάποιο τρόπο στην ανάπτυξη όσον αφορά θέση εργασίας. Υπάρχουν στοιχεία. Όχι. Α, βλέπω να κουνάτε το κεφάλι. Ε, βλέπω η απάντηση είναι αυτή. Δεν έχουμε. Ε δεν έχουμε αυτό το μέτρο αξιολόγηση, θα ήταν ε, σημαντικό να γνωρίζουμε. Για στόχους περιβαλλοντικούς υπάρχουν προγράμματα στον τομέα του περιβάλλοντος. Πάνω χάρη, ε, εξυγίανση, καθαρισμός διαφόρων βιομηχανικών περιοχών, μικρά έργα αν υπάρχουν. Θέσεις εργασίας, για να ξέρουμε και στον τομέα του περιβάλλοντος αν έχουμε κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νοβάκουφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Το θέμα είναι ύψη τη σημασία. Βέβαια, βλέποντα την παρουσία στην αίθουσα, θα θεωρούσε κανείς ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Ξέρω ότι αυτέ οι πράξει δημόσιο ιδιωτικού τομέα είναι από τις βασικές δυνατότητες που έχουν οι εθνικές αρχές και οι τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο επενδύσεων για τα κρίσιμα έργα τους. Μεγάλο το καθήκον που έχουν μπροστά μας, μεγάλο το έργο μας, έχοντας την έκθεση. Ποιο είναι αυτό? Να μεταφράσουμε αυτά που λέει έκθεση σε εύληπτη γλώσσα, κατανοητή για όλους τους πολίτες ή τουλάχιστον τους πολίτες που είναι υπεύθυνοι για ανάπτυξη διαφόρων έργων και προγραμμάτων στις χώρες να ξέρουν ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές, πώς μπορούν να μάθουν από τα μαθήματα που αναφέρονται στο έντυπο. Αυτό είναι καθήκον των μέλων, μελών της Επιτροπής. Υπέχουμε καθήκον να εξηγήσουμε το πώς χρηματοδοτεί και λειτουργεί η Ένωση και πώς μπορούν να προσελκύσουν τους ιδιωτικούς επενδυτές και να έχουν και την υποστήριξη της Ενώσεως. Νομίζω δεν είναι παράξενο, δεν είναι άξιο απορίας το ότι όσους πόρους και αν έχουν το δημόσιο τομέα, πάντα θα υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προσελκύσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια, χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές. Λειτουργεί το σχέδιο του Juncker ένα ποσό από το δημόσιο τομέα και να έχουμε στο βαθμό του δυνατού από τον ιδιωτικό τομέα για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα ε, για τους πολίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπηρεσία σας για την έρευνα που διεξήγαγε. Στέλνουμε τα καλύτερα μηνύματα, τα καλύτερα μαθήματα και θα τα προωθήσουμε σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων και έργων τουλάχιστον στο, στην εκλογική μου περιφέρεια, στη δική μου χώρα. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να θέσω κι εγώ μια ερώτηση. Αναφέρεται μερικές φορές τα κράτη-μέλη στα οποία έχουμε το μεγαλύτερο επίπεδο της χρήσης του PPP σαν εργαλείο για οικονομική διαχείριση και υλοποίηση των διαφόρων έργων. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ οικονομικής αναπτύξεως των περιοχών στις οποίες έχουμε αυτά τα προγράμματα PPP, εκεί που έχουμε υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής επένδυσης ή εκεί που χρειάζονται οι επενδύσεις και έχουν χαμελή, μικρότερη οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε κάποια στοιχεία. Διότι σε πολλές περιπτώσεις όπως εγώ είχα προτείνει το PPP για κάποια επενδυτικά σχέδια σαν επιλογή. Κυρίως οι περιφερειακές αρχές και η τοπική αυτοδιοίκηση ανταποκρίνονται λέγοντας ότι αυτή το εγχείρημα είναι πολύ δαπανηρό και δεν κάνει για όλους. Άρα αυτή είναι η ερώτησή μου. Υπάρχει σχέση. Κάποια σχετικά σχόλια πάνω σε αυτό θα σας παρακαλούσα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα σημεία ερωτήσει Να απαντήσω καταρχάς για μεσαίου μεγέθους PPP. Ε, τα περισσότερα PPP συνεπάγονται μεγάλες επενδύσεις για υποδομές και κυρίως μεγάλες ε, εταιρείε. Σε κάποιες περιπτώσεις στη Γερμανία έχουμε την αγορά των PPP που είναι πια ανεπτυγμένη σε περιφερειακό επίπεδο. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν και πολύ μάλιστα στις αγορές PPP. Δεν έχουμε στοιχεία όσον αφορά το αριθμό θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Δεν ήταν αυτός άλλωστε ο στόχος της εκθέσεως. Δεν εστιάστηκε πάνω σε αυτό, αλλά είμαι σίγουρη ότι πιθανότατα στη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο για ολοκληρωμένα έργα θα πρέπει να έχουν τέτοιου είδου στοιχεία. Δεύτερο, ποια η σχέση μεταξύ περιφερειακής αναπτύξεως και της χρήσεως των PPP και πόσο ανεπτυγμένοι θεσμοί και πόσο χρησιμοποιούνται τα PPP. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τι παρατηρήσαμε. Ακόμα και στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί πολύ το μοντέλο των PPP για να χρησιμοποιεί τα χρήματα των Ευρωπαϊκών διαθετικών ταμείων, η όλη προσπάθεια γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει τι περιοχέ, τι περιφέρειε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα. Το ίδιο ισχύει για την Πολωνία και για την Κροατία. Εξαρτάται κατά πολύ από την τεχνογνωσία που υπάρχει σε κάθε περιοχή και τη διαθέσιμη υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. πραγματικά πρέπει να πω ότι λυπούμεθα που οι συνάδελφοί μας απουσιάζουν, που δεν είναι εδώ να σας ακούσουν και να ακούσουν εξηγήσεις. Έχουμε όμως την έκθεση, έχει διανεμηθεί. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τους πω να απευθύνουν τις ερωτήσεις στην ομάδα που ετοίμασε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και τη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση επ' αυτού. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση πρωτοβουλίας που ετοίμασε ο συνάδελφος Αντρέη Νουβάκοφ πολιτική συνοχής προώθησης βοηώσιμων μεταφορών και κατάργηση των συμφορήσεων σε βασικές υποδομές δικτύων. Άρθρο 9.7 του κανονισμού του σχετικού. Ο λόγος στον κύριο Νοβάκουφ για να παρουσιάσει την θέση του επί της εκθέσεως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μου δίνει το λόγο. Τιμή μου, διότι για πρώτη φορά στην καριέρα μου εδώ αντιπροσωπεύω το 50% των μελών της Επιτροπής τεράστια ευθύνη. Πρέπει να το πω αυτό, να το παραδεχτώ. Εκτός της Προέδρου, εκτός της Προέδρου. Η Πρόεδρος εξαιρείται και εκτός του περίπλοκου τίτλου της εκθέσεως θα κάνω ό,τι μπορώ να σας εξηγήσω. Φαίνεται ότι είμαστε περισσότερα μέλη της Επιτροπής εδώ, δεν πρόσεξα. Λοιπόν, αφήσουμε εκτός τον πολύ περίπλοκο τίτλο της εκθέσεως να σας δώσω εγώ μια σύντομη παρουσίαση γιατί είναι σημαντικό το θέμα και γιατί ανέλαβα την πρωτοβουλία να επεξεργαστώ το θέμα. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια στην Ήπεθρο της Βουλγαρίας. Ε, λοιπόν, πιο φαρδής δρόμος και, και πιο γρήγορο τρένο σημαίνει καλύτερη ζωή. Μπορείς να πας τη δουλειά σου εγκαίρος, σου παραδίδουν τα προϊόντα εγκαίρος, οπότε η οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να μεγαλώσει καλύτερα, μπορεί να εξαρτηθεί καλύτερα από μια καλύτερη υποδομή, οδικό δίκτυο, καλύτερε υποδομέ. Άρα έχει μεγαλύτερε πιθανότητε, αν είναι καλύτερο το δίκτυο, να μην έχει και ατύχημα στον δρόμο. Διότι το τροχαίο ατύχημα είναι συνάρτηση του, ε, της ποιότητας του οδοστρώματος. Λοιπόν, οι μεταφορές επηρεάζουν τη ζωή όλων πιθανότατα. Κάθε μέλος της κοινωνίας. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Αυτές οι υποδομέ επηρεάζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η προσέγγιση μα στις μεταφορές δεν είναι ακόμα ένας τομέας πολιτικής, όχι. Είναι ένα δείγμα του πώς αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξη της ενώσεώς μας. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο. Προετοίμασα κάποια στοιχεία να σας παρουσιάσω. Δεν θέλω να αναφέρω τα στοιχεία, αλλά ακόμα και τα μισά από αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά πιστικά. Θα πιστούν όλοι που είναι πιο ε, διστακτικοί όσον αφορά τη σημασία που έχει το τομέα των μεταφορών. Είναι καλό που η Ένωση προετοίμησε, μάλλον προετοίμασε το δίκτυο TNT, το διευρωπαϊκό δίκτυο. Αν αναπτύξουμε το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών μέχρι το 2030, θα δώσουμε στους πολίτες 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 10 εκατομμύρια περισσότερες οικογένειες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να καλύψουν ανάγκες. 10 εκατομμύρια οικογένειες. Εάν δεν το κάνουμε, το αντίθετο δηλαδή, θα χάσουμε σχεδόν 2% του ΑΕΠ που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Θα χάσουμε 2% ανάπτυξης, τουλάχιστον. Σε ποσό είναι περίπου μισό τρεις. Τεράστια ποσά, εάν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Η έκθεσή μου θα εστιάζεται βέβαια επί των επιτευχθέντων από πλευρά μα. Πόσο αποτελεσματικέ ήταν οι επενδύσει και οι πρωτοβουλίε μα. Όμω θα δώσω όλη μου την ενέργεια και θα εστιαστώ και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να εφαρμόσω τις ιδέες μου που θα αφορούν οι ιδέες μου το μέλλον των επενδύσεων για τι μεταφορέ. Ποια θα έπρεπε να είναι η μορφή του στο μέλλον, διότι βλέπω κάποια ανησυχητικά σημάδια τελευταία χρησιμοποιήστε περισσότερα από τα χρήματα συνοχή. χρησιμοποιήστε τα, διοχετεύστε τα στο ΣΕΦ ή κάποιε άλλε ιδέες. Αυτό δημιουργεί, πώ να το πω, ε, μη προβλεψιμότητα, αστάθεια για τα κράτη-μέλη. Προσχεδιάζουν τη συμπεριφορά τους και επενδύσεις για κρίσιμα έργα και όχι σωστά δεν πρέπει να γίνεται αγώνας μεταξύ των διαφόρων φορέων τοπικών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων της Ένωσης. Εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκές οικογένειες, τη μοίρα τους. Άρα, πρέπει να είμαστε όσο πιο υπεύθυνοι γίνεται όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Επί του παρόντος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορούμε να χρηματοδοτούμε μέχρι το 1 τρίτο όλων των έργων των επιλέξιμων όσον αφορά το μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπης. Τα άλλα έργα είναι επιλέξιμα με καλούς δείκτες, αλλά δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να τα πραγματοποιήσουμε. Αν έχει προτεραιότητα το μέσο των μεταφορών για μας, τότε θα πρέπει να έχει προτεραιότητα το μέσο και στον προπολογισμό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Όμως, Νομίζω ότι οι έρευνε που έγιναν σύμφωνα στα πλαίσια του ΕΣΥΦ θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. Διότι οι δήμαρχοί μας, οι πολίτες μας, το αξίζουν και περιμένουν από μας να δώσουμε τα σωστά αποτελέσματα. Άρα, έχουμε κάποια βασικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν ότι μπορούν να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Πολύ λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Άρα, λιγότεροι τραυματίες, λιγότεροι θάνατοι λόγω ε, τροχαίων δυστυχημάτων, λόγω κακού οδοστρώματος. Παρέχουμε ένα καλό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αναπτυχθούν, διότι κάθε μία από αυτές, και εδώ ανοίγω παρένθεση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και παρέχουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των θέσεων εργασίας στην Ένωση. Κλείνω παρένθεση. Όλες λοιπόν οι επιχειρήσεις χρειάζονται καλές υποδομές, ούτω ώστε να πουλούν περισσότερα προϊόντα, να παρέχουν περισσότερες ε, υπηρεσίες. Σχεδόν κάθε πτυχή των πολιτικών μας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη, η ασφάλεια των δρόμων, ακόμα και εκπαίδευση και καινοτομία χρειάζονται μια καλή μεταφορική υποδομή. Και να πω κάτι που δεν είναι πολύ δημοφιλές. Πρόσφατα, σε διάφορες διασκέψεις, συνέδρια, οι περισσότεροι λένε ότι σε λίγα χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε οδηγούς διότι θα πετάνε, λέει ο μιλητής, τα αυτοκίνητα μόνο τους. Ε, δεν θα χρειαζόμαστε τρένα, θα έχουμε αεροσκάφη άνευ κυβερνήτου, θα έχουμε μια μη επανδρομένα επτάμενα οχήματα drones που θα παραδίδουν τρόφιμα. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα συστήματα. Ίσως εδώ να είμαι πιο συντηρητικό και παραδοσιακός. Ανεξάρτητα από την ψηφιοποίηση της ζωής μας, τα επόμενα έτη, και σημειώστε το αυτό, πάντα θα χρειαζόμαστε μεγαλύτερα λιμάνια, ευρύτερους δρόμους και ταχύτερα τρένα, διότι ζούμε σε έναν υλικό κόσμο. Άρα δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προτεραιότητά μας για επενδύσεις στις μεταφορές. Μάθαμε καλά από τα μαθήματα των τελευταίων ετών που πρέπει να βελτιωθούμε. Έχουμε κάποια παραδείγματα κυρίως όσον αφορά τις συμφορήσεις. Κάποια κράτη-μέλη αλυσιδωτά επενδύουν στον ίδιο μεταφορικό διάδρομο. Και η τελευταία χώρα που είναι στο τέλος του διαδρόμου δεν θεωρεί ότι αυτό είναι προτεραιότητα και δεν επενδύει. Άρα η υπόλοιπη επένδυση δεν έχει νόημα. Δεν θα χρησιμοποιηθεί. αν έχει ένα τρένο μπορεί να πάει 300 χιλιόμετρα την ώρα και περνάει, διατρέχει τα πρώτα τέσσερα κράτη-μέλη. Και όταν το τρένο πρέπει να φτάσει στην τελευταία χώρα και πρέπει να πάει με 60 χιλιόμετρα την ώρα, άρα δεν έχει νόημα να τρέχει πιο γρήγορα πριν. Δεν είναι αποτελεσματικό όσο θα μπορούσε το τρένο. Άρα αυτό πρέπει να το σταματήσουμε, να το εμποδίσουμε, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα. Και αυτό δεν γίνεται με το απόθεμα το οποίο έχουμε. Είχαμε υποσχεθεί στα κράτη-μέλη που θα έχουν απόθεμα βάση επιδόσεων για κάποιους λόγους. Και περιμένουν να το τηρήσουμε, να αλλάξουμε τους κανόνες πριν το τέλος του παιχνιδιού. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε τους στόχους μας και να πετύχουν καλά αποτελέσματα. Οι εταίροι μας από τα κράτη-μέλη αξίζουν προβλεψιμότητα, διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα κρατη και τα θέματα αυτά, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Οποιαδήποτε νέα κατανομή των χρημάτων πρέπει να εξεταστεί λίγους μήνες πριν έχουμε το νέο κανονισμό, πριν γίνει αξιολόγηση όσον αφορά τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στην αρχή της θητείας. Οι δεμοί, τουλάχιστον αυτοί που έχουν εκλεγεί, θα είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λογοδοτήσουν στο τέλος της θητείας. Γιατί κάναμε αυτό που κάναμε, τι πετύχαμε. Και όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, θα ήθελα να πάω σε αυτούς που με ψήφισαν και στο κόμμα μου και να μπορέσω να τους πω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ούτω ώστε να δώσω αυτό που τους αξίζει. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που συλλέγει λόγω ιδεών και αξιών και συναθρίζει τα κράτη-μέλη. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πίσω από τις λέξεις, τη σημαία και τον ύμνο υπάρχει ισχυρή πολιτική που παρέχει πόρους ούτως ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να γίνουν πλουσιότερα και να βελτιωθεί και η ζωή των λαών, η καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτά και ευχαριστώ οι σκιώδες εισηγητές. Ο κ. Πίκουλα είναι ο πρώτος, έχει το λόγο. Chair, I'll continue in my own language. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα αυτό το ζήτημα και να προετοιμάσουμε τις εργασίες μας, ε, τις μελλοντικέ για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Οι υποδομέ των μεταφορών είναι εξαιρετικά σημαντικέ για όλου του πολίτε μα και η Λευκή Βίβλο ανέφερε ότι η υποστήριξη τη ε, πολιτική συνοχή θα πρέπει να εστιαστεί στι βιώσιμε μορφέ των μεταφορών. Και από εκεί και μετά ε, αναφερόταν εκεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις συμφορήσεις, όλα τα bottlenecks, όπως αναφέρεται και στον 11ο στόχο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο στο 2020. Εάν λοιπόν αναφερθούμε ειδικότερα στο ζήτημα των εφιών μεταφορών, αλλά και των καθαρών, των clean μορφών μεταφοράς, ε, ειδικότερα στο πλαίσιο της αστικής κινητικότητας, τότε σίγουρα θα χρειαστεί υποστήριξη τόσο από το Ταμείο Συνοχής όσο και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε επενδύσεις οι οποίες θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο μέσα στην τρέχουσα ε, περίοδο χρηματοδότησης. Και ε, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική σχεδίαση αυτών των επενδύσεων και αυτό αναφέρθηκε ήδη ότι δηλαδή θα πρέπει να υιοθετηθεί από την πλευρά όλων των κρατών μελών ένα γενικό σχέδιο σε ό,τι αφορά τις μεταφορές τους έτσι ώστε από εκεί και μετά να προβλέπονται συγκεκριμένα έργα ε, τα οποία με την από την πλευρά τους θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων. Για παράδειγμα, τα 750 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, επενδύθηκαν ε, στην Τσεχία στο συνδρομικό δίκτυο θα έπρεπε να λάβουν περαιτέρω συνέχεια. Τα 30 εκατομμύρια που επενδύθηκαν στην Ουγγαρία στο συνδρομικό δίκτυο ε, αλλά και τα 17.000 ε, ε, τα 17 συγγνώμη, εκατομμύρια ευρώ τα οποία επενδύθηκαν στο συνδρομικό δίκτυο της Πολωνίας ήταν εξίσου σημαντικά. Αλλά θα πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω αυτά τα δίκτυα. Εγώ για παράδειγμα κατάγομαι από την Ουγγαρία και τα προβλήματα ε, στις μεταφορές παραμένουν εστιασμένα στο μεγαλύτερο βαθμό στις συνδρομικές ε, μεταφορές. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε παραπέρα εδώ. Ε, ίσως λοιπόν η πολιτική συνοχή θα έπρεπε να δώσει περαιτέρω έμφαση σε αυτούς τους θεματικούς στόχους, αλλά επιτρέποντας προφανώς και τα απαραίτητα ε, περιθώρια ευελιξίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες ε, των περιφερειών. Θα πρέπει για παράδειγμα πάντοτε να έχουμε κατά νου κατά πόσο έχουμε να κάνουμε μια αστική ή με μια υπαίθρια περιοχή. Ή θα πρέπει να, κάνουμε, να, να, να έχουμε πάντα κατά νου να έχουμε να κάνουμε μια ανεπτυγμένη ή μια αστερούσα περιοχή. Επίση θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα και τι οι γεωγραφικέ ιδιαιτερότητε των περιοχών. Για παράδειγμα, εδώ αναφέρομαι στις ε, βόρειες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, όπου η πυκνότητα, δηλαδή η πληθυσμιακή, είναι πολύ χαμηλή. Ε, ακόμα και το ζήτημα, για παράδειγμα, της, των απομονωμένων κοινοτήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, των απομονωμένων περιοχών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει ω παράγοντε να λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε ε, το δίκτυο μεταφορών μας επιτρέποντας ακριβώς και την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων όχι μόνο σε κάποια μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο σύνολό τη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαρμέλ Τέρμπορκ, ε, επόμενος σκιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο και έχασα το πρώτο τμήμα της ε, παρέμβασης του κύριου Νόβακοφ, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα το ξανασυζητήσουμε. Όταν μιλάμε για βιώσιμες μεταφορές και την ε, ε, εξάλληψη των συμφορήσεων, ε, έχουμε μέντε το, την διευκόλυνση ιδέοντας στην Ευρώπη, αλλά και το ΕΦΣΙ, το σχέδιο Juncker. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συνέργειες ανάμεσα στο ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ε, συνδέοντα την Ευρώπη, ώστε να συνδυάσουμε και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα ευρωπαϊκά project που θα δημιουργήσουν περισσότερη προστιθέμενη αξία. Στι μεταφορέ θα πρέπει να θυμόμαστε ε, και την Επιτροπή Μεταφορών. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με ευρωπαϊκά χρήματα ένα διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και χρειαζόμαστε πολλά λεφτά γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να βρούμε όλα τα ευρωπαϊκά χρήματα που είναι απαραίτητα όχι μόνο για να χρηματοδοτηθούν οι κύριοι διάδρομοι, αλλά και ολόκληρο το δίκτυο. Γι' αυτό θέλω να κάνω μια ανέκκληση για τη συμπερίληψη των ε, μικρών project ε, διασυνοριακών υποδομών γιατί έχουμε και μία νέα γενιά προγραμμάτων Interreg μετά το 2020, γιατί νομίζω πως ορισμένα από τα χρήματα στο τομείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα επενδύσουμε σε project που είναι πραγματικά απαραίτητα για να βελτιωθεί και η διασυνοριακή συνεργασία στις ε, συνοριακές περιοχές. Όταν μιλάμε για επενδύσεις υποδομών, κατά τη γνώμη μου πρέπει να εστιάσουμε στα εξή σημεία. Πρώτον, την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή να ευνοήσουμε τρόπους μεταφορών πιο φιλικούς προς το περιβάλλον, καθώς και να ε, πληρώνει ο χρήστης ε, τους, ε, τα είδη μεταφορών που χρησιμοποιεί, όπως ας πούμε τα διόδια για τις οδικές μεταφορές. Θα πρέπει να μείνουμε σε αυτή την αρχή που αποτελεί και τμήμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι και το κομμάτι του πακέτου για την κινητικότητα, δηλαδή χρέωση το, της χρήσης των δρόμων μέσω της Ευρωβινιέτας. Έπειτα έχουμε διάφορα ε, δίκτυα τώρα εθνικά, ε, θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Συχνά τα διασυνοριακά project θεωρούνται λιγότερο σημαντικά από τις εθνικές αρχές, όμως υπάρχει μια πραγματική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται όταν υλοποιούνται αυτά τα έργα. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στις συμφορήσει και στου αδύναμου κρίκου γιατί έτσι μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη των συνολικών περιοχών της Ευρώπης. Η τρίτη μου αρχή, που είναι επίσης νομίζω πολύ σημαντική, είναι να το χρησιμοποιήσεις, αλλιώς θα το χάσεις. Αυτό εισήχθη μέσω της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη και ορίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το στόχο για τον οποίο είχε προβλεφθεί και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν το καταφέρει αυτό το κράτος μέλος, τότε χάνει αυτή την ε, χρηματοδότηση αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα αλλά και ε, τους χρόνους ε, κατασκευής των έργων. Προσβλέπω συνεργασία μου με τον κύριο Νοβακόφ για αυτή την ε, έκθεση. Πρέπει όντως να δρομολογήσουμε πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση και πιο στοχευμένη χρηματοδότηση για τις μεταφορές ώστε να έχουμε και προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Βαλίνα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Νταμάτο. Κύριε Ρόπε, όχι. Ωραία, η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τι έχω, 20 λεπτά? Όχι, δεν μου αφήνετε. Καντάξει. Eh, Αυτή η έκθεση μιλά για μια σημαντική ε, πτυχή των πολιτικών της Ένωσης, δηλαδή βιώσιμη ανάπτυξη οδικών δικτύων και δικτύων μεταφοράς, μεταφορών. Αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά για την επίτευξη μια σειρά στόχων. Α πούμε, οικονομία με χαμηλό ή και μηδενικό δίκτυο πομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανάγκη μείωση ε, του διαφοράς μεταξύ αστικών κέντρων και ε, περιοχών της υπαίθρου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι η συνεργία ανάμεσα στο Ταμείο Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης ε, και το ΕΦΣΙ και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα διευθυντικά ταμεία, αν και δεν ξέρουμε ακόμα πόσα θα είναι τα χρήματα που θα μείνουν στην πολιτική συνοχή ε, για τις μεταφορές. Το τόνισαν αυτό και άλλοι συνάδελφοι. Στη χώρα μου, στην Νότια Ιταλία, πάντοτε αυτές οι περιφέρειες που περισσότερο θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα διευθυντικά ταμεία είναι εκεί και έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εκεί όπου ενώ, έχουμε διάφορους πόρους για διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα γιατί οι βιώσιμες μεταφορές, ή τοπικέ και περιφερειακε αρχες αρχές έχουν υποβάλει μόνο ένα-δύο project από το 2014 είναι μια κατάσταση πραγματικά ανησυχητική γιατί ο προπολογισμό στο ε, Ταμείο Συνοχή είναι 20 δι. Καλά κάνουμε λοιπόν και επιμένουμε για τη συνεργασία. Για να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα, μπορεί εμεί να αποφασίσουμε να μεδίσουμε στι ηλεκτρονικέ μεταφορέ, αλλά να δεν δώσουμε κίνητρα για τη χρήση και την παραγωγή ε, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αν δεν έχουμε την οικονομία της φόρτισης και δεν έχουμε την κατάλληλη τότε δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά. Να θυμίσω ότι αυτός ο στόχος ε, ε, ε, θέλει να βοηθήσει στην κινητικότητα ανθρώπων και ε, εμπορευμάτων μέσω της ισορροπίας και με τη χρήση ε, τρόπων μεταφοράς που μολύνουν λιγότερο, να βελτιωθεί η κατάσταση περιβάλλοντος και οι όροι διαβίωσης. Αυτά συνδυάζονται με τη βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και των υπηρεσιών που, που, που, που παρέχονται, καθώς και την ενίσχυση των λιμένων, καθώς και της σχετικής επιμελητίας. Όμως τα κράτη-μέλη μεμονωμένα αντιμετωπίζουμε και συγκεκριμένα στην Ιταλία και στη Γαλλία, ε, προσκρούμε στην ε, βούληση να δημιουργηθεί αυτή η ταχεία ε, κυκλοφορία στη δρομική γραμμή το Ρήνο Λιών, ενώ υπάρχουν ε, ε, περιφέρειες οι οποίες δεν το επιθυμούν shift άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια χρηματοδότηση θα δοθεί στις συνδρομικές μεταφορές μικρής ε, εμβέλειας, ε, όχι μόνο στα τρένα μεγάλης ταχύτητας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα νέο τρόπο ε, κοινωνίας πάνω στο πρότυπο του εφιούς κράτους χωρίς να αφήσουμε όμως κανέναν πίσω. Ένα μοντέλο κοινωνίας όπου οι πολίτες ε, είναι ενημερωμένοι ε, και ξέρουν τα ωφέλη των νέων συστημάτων κινητικότητας ε, που στο, στόχο να έχουμε την οικοβιωσιμότητα για να βελτιωθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν και νέες θέσεις απασχόλησης. Στόχος μας είναι ως μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θεματικός στόχος 3 που αναθέσαμε και προηγουμένως θα πρέπει λοιπόν να, να συλλάβουμε μια συνολική εικόνα που θα ενθαρρύνει τη χρήση των δημοσίων μέσων μεταφοράς για να μειώνουμε τις εκπομπές, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, αλλά και να διευκολύνουμε την μικροοικονομία των ε, αστικών κέντρων. Thank you. As I do not see any other wishes for, Μάλιστα, ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Δεν βλέπω. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζιούκ αν τον προ, πρόφερα σωστά το όνομά σας, με συγχωρείτε αν έκανα λάθος. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG Regio. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ρόμπερτ Σφίτσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτής ε, της ε, έκθεσης της Επιτροπής Μεταφορών και είμαστε της ίδιας άποψης ότι δηλαδή πρέπει να βρεθεί η δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων ε, μέσων χρηματοδότησης της Κομισιόν και υπάρχει κοινό προβληματισμός ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες για την ώρα για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια έναν συνδυασμό όντως αυτών των πόρων αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλα όσα ακούσαμε για τις τοπικές ε, αστικές μεταφορές, τις αυτοματοποιημένες μεταφορές, όπως είπατε, σχεδόν αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής και δεν μπορούμε να γνώουμε ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες. Χρειάζεται παρέμβαση και συντονισμός για το πώς θα γίνουν όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να συντονίσουμε ποιος ασχολείται με τι στο καλύτερο επίπεδο και στο καλύτερο συντονισμένο επίπεδο. Η διασυνοριακή διάσταση είναι βεβαίως πολύ σημαντική. Ε, ακριβώς ε, εδώ είναι που συνεχίζουν τα κράτη-μέλη να ασχολούνται, να βρίσκουν τη διαλειτουργικότητα και τα απλούστερα ευρωπαϊκά συστήματα μεταφορών, ώστε να συμβάλλουμε και περισσότερο στην ανάπτυξη νέας αγοράς. Ενθαρρύνουμε αυτού του είδους τις επένδυσεις. Which was mentioned is was the new feature, the extended conditionality for having a transport plan for. Έχουμε ένα σχέδιο μεταφορών για να μπορέ... που χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μέσω της πολιτικής συνοχής. Αυτή ήταν μια μεγάλη πρόκληση και για μας και για τα κράτη-μέλη και για τις περιφέρειες. Αλλά τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και έκαναν την απαραίτητο στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να υπάρξει αυτή η στέρη βάση για τις επενδύσεις της μεταφορές. Είναι ένα καλό παράδειγμα από τις τρέχουσες προοπτικές και πρέπει να δούμε πώς περαιτέρω θα το ενισχύσουμε αυτό. Θέλουμε να προσφέρουμε την υποστήριξή μας ε, στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νόβακοφ, θέλετε να ολοκληρώσετε εσεί τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, τιμότητα και, την ε, προσέγγιση των συναδέλφων, των σκιωδών εισηγητών, αλλά και του εκπροσώπου της Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι η αρχική συζήτηση ήταν καλή αρχή. Έχουμε δημιουργήσει ένα καλό περιβάλλον, ώστε τον Μάιο, ε, γενικά την άνοιξη του χρόνου, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτά από την πλευρά μου μέχρι στιγμής. thank you very Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι περιμένουμε το σχέδιο εκθεσή σα για το Φεβράριο. Θα είμαστε λοιπόν ε, εντός των προθεσμιών και τώρα... Έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση της ημερησίας μας διάταξης. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Τις εγκρίνεται, δεν υπάρχουν σχόλια. Ωραία, εγκρίνονται. Any other business? Υπάρχει κάτι να συζητήσουμε στα διάφορα. Όχι. Να θυμίσω ότι η επόμενη μας συνεδρίαση θα είναι μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 5. Η τακτική μας συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου. Και 25 Ιανουαρίου το πρωί. 24 Ιανουαρίου και 25. These are my, my announcements for the next meeting and um, may I ask to uh, may I thank to the interpreters for their support for today's meeting and uh, I uh, close the meeting of Regi Ευχαριστώ και τους διερμηνείς και εδώ λίγη η σημερινή μας συνεδρίαση.